Kolleginnen Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε τόσο πολύ άριθμοι παρά την ε, πρόσκληση που ήταν σχετικά πρόσφατη. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία μετά από αίτημα του Προέδρου του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά συζήτηση με τον, Ουκρανό Πρόεδρο, με τον Ουκρανό Πρόεδρο και σε ό,τι αφορά την ε, κατάσταση να λάβουμε μία απόφαση σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα αποφασίσει το Συμβούλου και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, αν θέλουμε να προλάβουμε την Ολομέλεια, να πάρει σήμερα απόφαση η Επιτροπή μας. Σε συνεργασία λοιπόν με την Επιτροπή ΙΝΤΑ ανακοινώσαμε ότι δεχόμαστε τη διαδικασία αυτή και αυτό θα αφορά μόνο τη συνάντησή μας και όχι το ψήφισμα το οποίο θα κληθούμε σε μετέπειτα χρονική στιγμή να καταρτήσουμε λόγω και του χρόνου που χρειάζονται οι εισηγητές. Συνένεση. Συνένεση προκειμένου λοιπόν να συνεχίσει η διαδικασία για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Και ο εισηγητής ε, Σάρις Βόλφσκι ήταν σύμφωνος με τη διαδικασία αυτή. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για το αίτημα αυτό. Συμφωνείτε με την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Ο κύριο Σόλτ ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ σύνθετη και δύσκολη ε, διαδικασία και εδώ καλούμαστε να εξαγάγουμε τα καθήκοντά μα. Ζητάω ε, σεβασμό σε ό,τι αφορά με όλο το σεβασμό προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κατά πόσο έχει νόημα στην παρούσα φάση με ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι διχασμένο και όπου επικρατούν πολλές και διαφορετικές καταστάσεις να συνεχίσουμε την διαδικασία επικύρωσης χωρίς να έχει γίνει η σχετική συζήτηση για το θέμα αυτό. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι είναι πολύ διαφορετικές οι απόψεις εδώ στην Επιτροπή μας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ενδεχομένως θα άξιζε να σκεφτούμε πρωτού να το σκεφτούμε αυτό άλλη μια φορά πριν κάνουμε την ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιο αντίθετο με το αίτημα αυτό, λέει ο πρόεδρο. Να ακούσουμε ποιο είναι κατά και μετά να αποφασίσουμε για την αναβολή ε, ενδεχομένως της, ε, του σημείου αυτού της ημερήσια Ποιος είναι λοιπόν κατά. Πώ είναι κατά τη ε, του κ. Σόλτ. Απορρίπτεται λοιπόν το αίτημα του κυρίου Σόλτ. Και περνάμε λοιπόν έτσι στο 3 της ημερής διάταξη. διάταξης. μικροφώνου. Μπορούμε αυτό να καταγραφεί επισήμως, να ζητήσουμε να καταγραφεί αυτό επισήμως. Κύριε Πρόεδρε, η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ γιατί είναι καταλαβαίνετε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Δεν το είχατε ζητήσει, λέει ο Πρόεδρος, και είναι πολύ αργά και πολύ λυπάμαι. Αργήσατε. Το ζητώ εγώ. leave the room when you ask. Παρακαλώ να εξέλθω τις αιθούσεις, λέει ο Πρόεδρος. Uh, here was an amendment to change the order έγινε έτοιμα να αλλάξει η σειρά της ημερήσιας διάταξης. Κάποιος μίλησε κατά και ψηφίσαμε. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία που ακολουθείται και στην Ολομέλεια. Ένας μιλάει υπέρ, ένας μιλάει κατά και μετά γίνεται ψηφοφορία. Δεν ζητήθηκε προηγουμένως, αλλά όταν φύγετε από την αίθουσα μπορεί να κάνουμε την κοινωνική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίζεται υπέρ του κυρίου Σόλτς ή κατά του κυρίου Σόλτς. Αυτή είναι η τροπολογία επί της οποίας ψηφίζουμε. Η τροπολογία που προτείνει ο κύριος Σόλτς. So, there are still some people who have not voted yet. Δεν έχουν ψηφίσει όλοι ακόμα. And then use your American Express. Χρησιμοποιήστε την πιστοτική σας κάρτα, λέει ο Πρόεδρος, άμα δεν έχετε κάρτα ψηφοφορίας. Okay, we will record that. So, the vote is... Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ψηφοφορία. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 9, 48 κατά, 2 αποχές. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την ατζέντα όσο προβλέπετε. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση. Αν δεν είναι έκθεση, διορθώνει ο πρόεδρος. Συνένεση. Και ο εισηγητής θέλει να πάρει το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, υποβάλλω προς ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφενό και της Ουκρανίας αφετέρου. Για δύο λόγους. Θέλουμε να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και αλληλεγγύη με την ευρωπαϊκή επιλογή που έχει κάνει η Ουκρανία, που είναι πολύ χειρή και πολύ τολμηρή σε όλα τα στρώματα της Ουκρανικής κοινωνίας. Επίσης, για συμβολικούς λόγους θέλουμε ε, την επικύρωση αυτή που αν πούμε σήμερα ναι και υπερψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε στην Ολομέλεια ώστε παράλληλα με τη Βίρχοβνα Ράντα δηλαδή την Ουκρανική Βουλή να κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία σύνδεσης. Άλλωστε συνταγματικά είναι απόλυτα ικανή η Βίρχοβνα Ράντα, η Ουκρανική Βουλή, να κυρώσει αυτή τη συμφωνία σύνδεσης όπως θα κάνουμε και εμεί σήμερα και η Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα. Σα καλώ λοιπόν να εγκρίνουμε αυτό το σύντομο νομοθετικό ψήφισμα που λέει στο σημείο 1 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τη συνένεση για τη σύναψη της συμφωνίας. Αυτά, ευχαριστώ. Ο κύριος Σούμπελ, που είναι αρμόδιος της εξωτερικής υπηρεσίας, ε, χαίρομαι για την πρόταση αυτή να ε, γίνει ταυτόχρονη κύρωση από τη Βίρχο Βαναράδα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Συμφωνία, γιατί είναι κρίσιμη στιγμή για την ε, Ουκρανία και μια τέτοια απόφαση θα είναι συμβολικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τα, τα, τις εμπορικές προτιμήσεις ήδη έχουν φέρει αποτελέσματα και 14% αύξηση των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι δίνει δίνουμε την ευκαιρία στην Ουκρανία να δείξει τις εξαγωγικές της ε, δυνατότητες. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα μεγαλύτερα ωφέλη της συμφωνίας και για τις δύο πλευρές. Όπως ξέρετε κύριε Πρόεδρε και αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία στη διάρκεια της, ε, του έτους ε, είχαν συνομιλήσει με την Ρωσία για να εξεταστούν τα οικονομικά ε, αποτελέσματα της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης ε, και της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου για να αντιμετωπιστούν κάποιες ανησυχίες και να βρεθούν λύσεις. Μία πρώτη τριμερής υπουργική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε στις 11 Ιουλίου. Η διαδικασία κύρωσης από την Ουκρανική πλευρά συνεχίζεται όπως είχε προγραμματιστεί. Βέβαια χρειάζονται περαιτέρω συζητήσει ε, για να ε, διελευκανθεί ο αντίκτυπο σε Ουκρανού και Ρώσου της εφαρμογή της συμφωνίας. Και μάλιστα την ε, Παρασκευή θα γίνει νέα υπουργική διάσκεψη με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Ντεχούχτ και με τους ομολόγους του από την Ουκρανική και Ρωσική πλευρά. Δίνονται νέες ευκαιρίες και είναι σημαντικό βήμα στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Ουκρανία στη διαδικασία μεταμόρφωσης προκειμένου να, γίνει μια σταθερή και ευημερούσα δημοκρατία. Και εύχομαι καλή τύχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία κύρωση τη συμφωνία αυτή. Ο κύριος Πλέγκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ως να εκλεγείς πρώτος, πρώτος αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, για την Ουκρανία στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Θα ήθελα να στηρίξω το αίτημα του κύριο Σάριου Βόλσκι, ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να κυρώσουμε σήμερα αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να αποφανθεί Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Κάτι τέτοιο άλλωστε δείχνει την ισχυρή δέσμευση όλων των πολιτικών ομάδων να συνεχίσουμε να στέλνουμε θετικά μηνύματα προ την Ουκρανία, ιδιαίτερω στηρίζοντα την ευρωπαϊκή τη επιλογή. Και όταν ξεκινήσει μετά τον Νοέμβριο, ευελπιστούμε μετά τις εκλογέ η εφαρμογή τη συμφωνία, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους συναδέλφους ομολόγους μας Βίρχοφνα Ράντα για την εφαρμογή της συμφωνίας και για τις μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν όμως την εδαφική ακερότητα της Ουκρανίας. Ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Εγώ ως και ο θεωρώ ότι εμείς οι ευρωβουλευτές με θετική ψήφο της, του νομοθετικού αυτοψηφίσματος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δείξουμε ε, υποστήριξη για κάτι και όχι να δείξουμε αντίσταση απέναντι σε κάτι. Και η υπερψήφιση αυτής της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης ε, δείχνει πραγματικά μια υποστήριξη. Είναι σημαντική συμβολή προκειμένου να αρθούν κάποια διλήμματα για το μέλλον της Ουκρανίας. Δεν είναι ούτε θα έπρεπε να γίνει έρμεο ή υποτελής μιας πρώην ε, σοβιετικής περιοχής αλλά να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στήριξη αυτής της συμφωνίας σύνδεσης είναι σημαντικό μήνυμα προς την Ουκρανία, ότι τη βλέπουμε σαν εταίρο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και σημαντικές δυνατότητες να εγκρίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αν δεν γίνουν διευρύσεις στην ε- Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη πενταετία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Ουκρανικό λαό να συνεχίσει τις ενταξιακές του βλέψεις και να μην διαψευσει τις ενταξιακές του προοπτικές. Ευχαριστώ.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 παράδοση στην υποστήριξη της ε, ουκρανικές ε, ευρωατλαντικές προσδοκίες και την προσχώρηση της Ουκρανίας στην Ένωση μία μέρα των ημερών. Δεν θα σας εντυπωσιάζει λοιπόν για μένα ως συντονιστή και το σύνολο της αντιπροσωπείας μου στην ΑΦΕΤ ότι θέλουμε πολύ να βοηθήσουμε στην Ουκρανία, την Ουκρανία τη στιγμή που ρωσικά στρατεύματα εισβάλλουν ε, στην επικράτειά της και προσαρτούν την Κρυμαία. Θέλουμε να κάνουμε την μπορούμε να βοηθήσουμε τον ε, πρόεδρο Μποροσέγκο και τους ε, συναδέλφους του που αγωνίζονται με ρωσικά τάγκ στην επικράτειά τους όσο γίνεται πιο σύντομα. Και αν αυτό ε, γίνει πιο επιταχυμένα ώστε να συμβεί αυτό ταυτόχρονα με την επικύρωση από την Ράντα στο Κιέβο θα ήταν μια συμβολική χειρονομία ώστε να δείξουμε αλληλεγγύη με το λαό της Ουκρανίας και την κυβέρνησή τους αυτή τη στιγμή που τόσο το έχουν ανάγκη. Οπότε μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξη τη δική μου μας. Σας ευχαριστώ. Λέζινγκ. Οι βουλευτές της GUNGL θα καταψηφίσουν την επικύρωση της συμφωνίας εδώ, σήμερα. Ο συνάδελφος κύριος Σόλτς ανέφερε ήδη κάποια από τα επιχειρήματά μας τα οποία μας ε, οδηγούν στην καταψήφιση σίγουρα της πρότασης αυτής. Μία προϋπόθεση, μία από τις προϋποθέσεις θα έπρεπε να είναι η κοινωνική σταθεροποίηση στην, ε, και ισότητα στην Ουκρανία γιατί η συμφωνία όπως έχει σήμερα περιλαμβάνει πολλά σημεία με τα οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε συνεργασία σε θέματα ασύλου, πολιτικής ασύλου, ιδιαίτερως ε, η συνεργασία σε ό,τι αφορά θέματα της Frontex, οι αρχές του ελευθέρου εμπορίου οι οποίες κατοχυρώνονται εδώ στην συμφωνία αυτή είναι κάτι το οποίο απορρίπτουμε και δεν θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν και θα οδηγήσουν τον Ουκρανικό λαό σε ευημερία. Απορρίπτουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία αυτή γιατί αποτελεί μια προσέγγιση σε θέματα πολιτικής ασφαλείας και θεωρούμε ότι αυτή η συνεργασία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και εξαιρετικά αντιπαραγωγική σε μια ερνευτική τέτοια φάση και διαδικασία στην Ουκρανία, μια συνεργασία η οποία δυστυχώς ε, ήδη προκύπτει ε, στην αποστολή Αταλάντα και σε άλλα battle groups, σε άλλες ομάδες μάχης. Ε, θα καταψηφίσουμε λοιπόν αυτό το αίτημα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ο κ. Παμπάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η φιλελεύθερη, η ομάδα της Άλντε, θα υποστηρίσουν αυτό το νομοθετικό ψήφισμα για να επικριθεί η Συμφωνία Σύνδεσης. Το συζητήσαμε και το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα με διάφορες κυβερνήσεις ε, στο Κίεβο. Είναι λοιπόν κάτι το θετικό για την Ουκρανία, κάτι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να γίνει κατανοητό και στη Ρωσία ότι μια ανεξάρτητη, ευημερούσα και ε, ελεύθερη Ουκρανία είναι κάτι καλό για τη σταθερότητα όλη τη περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσουμε υπέρ. Ο κύριο Κάβερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι κατά του ψηφίσματο αυτό και θεωρώ ότι η χρονική συγκυρία είναι αποτροπιαστική. Η κατάσταση είναι... κλειδονίζεται για κεχηρία. χιλιάδε έχουν χάσει τη ζωή του στην Ουκρανία και ε, προκαλούμε τη Ρωσία σας παρακαλώ λοιπόν και καλό όλους σας να σκεφτείτε πάρα πολύ προσεκτικά όταν αύριο το πρωί κοιταχτείτε στον καθρέφτη όταν θα ξερίζεστε και θα βάθεστε μπορεί να δείτε ένα πρόσωπο που έχει προκαλέσει περαιτέρω από τραπιαστικές ε, ενέργειες από λόγω της ματαιότητας αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μέζεριτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρόλο που συμμεριζόμαστε Κάποιε ανησυχίε για μερικέ λεπτομέρειες συμφωνίας σύνδεση. Γενικώ είμαστε υπέρ και ανεπιφύλακτα της συμφωνίας. Οι πράσινοι θα την υπερψηφίσουν για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό είναι ο μοναδικός τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δείξουμε αποτελεσματικά την ελεγγύη μας προς την Ουκρανία. Γιατί η απόρριψη μια τέτοια συμφωνία που ζήτησε η Ουκρανική Βουλή θα ισοδυναμούσε με υπονόμευση της εσωτερικής ουκρανικής, πολιτικής. Και έτσι θα δημιουργήσουμε περαιτέρω αναταραχές στην Ουκρανία με μια απόρριψη. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε όσο γίνεται. Ας μην ξεχνούμε επίσης ότι έτσι δεν θα λυθεί το θέμα ασφάλειας και τα στρατιωτικά ζητήματα στην Ουκρανία, γιατί είναι επισφαλής ακόμη η χειρία και σίγουρα εμπορικέ συμφωνίες δεν πρόκειται να αποκαταστήσουν την ασφάλεια. Γι' αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε και μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Ο κύριος Κόρβιν Μίκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Στην αρχή ανατρέψαμε τον κύριο Γιαννουκόβιτς, έπειτα έγιναν οι φασαρίες στο Μεϊντάν, σταθεροποιήθηκε μετά η κατάσταση στην Ουκρανία, έπειτα προκαλέσαμε την Ουκρανία να στραφεί κατά της Ρωσίας και τώρα αρνούμεθα να πωλήσουμε όπλα στην Ουκρανία. Αυτοί που το έκαναν είτε είναι πράκτορες του Πούτιν, είτε απλώς ηλίθιοι. Λυπούμε, αλλά το 1939 η Πολωνία δέχτηκε τις εγγυήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Άμεση επίθεση από τον Αδόλφο Χίτλερ. Σας παρακαλώ να μην κάνουμε πάλι το ίδιο λάθος. Κοιτάξτε στον καθρέφτη, όπως είπε ένας από τους προηγούμενους. Είστε Πολωνός ευβουλευτής, αν τα κατάλαβα. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να πω ότι το ΕΛΚ ε, υποστηρίζει την πρόταση του εισηγητού Σάριου Βόλσκ και θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους, όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, να μην ξεχνούν κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας ότι πολλοί άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να υλοποιηθεί αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέντα και επιτρέψτε μου μια προσωπική παρατήρηση. Νομίζω ότι να αποκλειστεί αυτή η συμφωνία ε, σε ό,τι αφορά την Ουκρανική λαό, το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει κατά πόσον θα υπερψηφίσει. Ο πρόεδρος, ο τρέχον, εκλέχθηκε για την ε, υπερψήφιση αυτής της συμφωνίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το καθοριστικό που πρέπει να δούμε. Η βία δεν ξεκινάει από την Ουκρανία, αλλά από τον ε, μεγάλο γείτονα της Ουκρανίας. Ο κύριος Γιαννουκόβιτς δεν ε, ε, τον διώξαμε, εγκατέλειψε την ε, θέση του. Και ο πρόεδρος ε, έχει νομιμοποιηθεί από άμεση εκλογή από τον λαό. Αυτή είναι η κατάσταση όσο έχει. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που ζητάει το λόγο και έτσι μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά κατευθείαν. Έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. Α, οι τροπολογίες. Να ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες, διορθώνει ο Πρόεδρος. Έχουμε την τροπολογία 1. Υπέρ. Hm? E Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ, κύριε Πρέντα. Μάλιστα. Τώρα είμαστε εντάξει. Δεν έχετε την κάρτα σας. Πέρα στις ψηφοφορίες λοιπόν για την τροπολογία 1. 8 υπέρ 49 κατά 4 αποχές. Και τώρα περνάμε λοιπόν στην τροπολογία περιθμών 2. Ηλεκτρονικά και πάλι ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 2. Abstimmung ist geschlossen. Ίδιο το αποτέλεσμα ή τουλάχιστον συγκρίσιμο. Και τώρα να ψηφίσουμε την πρόταση Σάριος Βολσκή. Ονομαστική κλίση. Έναρκτη τη ψηφοφορία. Γεια. Τένοκ μητιά. Και ο κύριο Τάνοκ που έχει ξεχάσει την κάρτα του ψηφίζει υπέρ. Πέρασε της ψηφοφορίας. 49 ψήφοι υπέρ, 8 κατά, 4 αποχές. Νομίζω ότι είναι, είναι συντριπτικό το αποτέλεσμα. Thus, Ukraine will lose, not new Russia. Ich äh, möchte hier zum Ausdruck bringen. Θα ήθελα να εκφράσω το εξή, λέει ο Πρόεδρος.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 Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ja, machen wir nächstes Mal. Das ist äh, pro forma. Jetzt Tagesordnungspunkt 4. Σημείο 4 της μερικής διάταξης έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον μεγάλο μουφτή της Αιγύπτου, ε, ο οποίος τυχαία βρίσκεται εδώ σήμερα και θεωρήσαμε ότι χρήσιμο κεφάλι μου θα ήταν να διεξαγάγουμε μια συζήτηση. Σε δύο λεπτά θα καταφτάσει. Luca, ha tutto a posto con la interpretazione 25. Colegas, vamos a... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσουμε ολόθερμα τον εξοχότατο δόκτωρα Σούκη Ισραήλ Σούκη Αλάμ που είναι καθηγητής νομολογίας στην Σχολή Σαρίας και Δικαίου του Πανεπιστημίου Αλτσάχαρ. Είναι ιδιαίτερη τιμή η παρουσία σας εδώ, εξοχότατε, γιατί είστε από τους σημαντικότερους εμπειρογνώμονες της μελέτης της Σαρίας και του Ισλαμικού Δικαίου. Και μάλιστα ξεκάθαρα δηλώσατε ότι όσοι χρησιμοποιούν το Ισλάμ ως άλοθη για την τρομοκρατία παραβιάζουν τις ανθρωπιστικές αρχές του ίδιου του Ισλάμ. Μιλήσαμε για, το, για την Αλκάιντα, ε, για το Ισλαμικό κράτος, αυτό το μεγάλο κακό. Είπατε... Είπατε και εσείς ότι πρόκειται για διαφθαρμένες ε, εξτρεμιστικές ομάδες, αιμοβόρες και αιμοδιψείς που παραβιάζουν και το Ισλάμ και τα ανθρωπιστικά δικαιώματα και συνιστούν απειλή για όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ιράκ ε, είναι η απειλή του Ισλαμικού κράτους για όλους τους ε, υπηκόους. Είτε είναι χριστιανοί, μουσουλμάνοι ή οποιασδήποτε άλλες ομολογίες θρησκείας. Πριν σας δώσω το λόγο εξοχότατε, θα ήθελα να λάβετε υπόψη τη βαθύτατη ανησυχία μας γιατί έχει γενικευθεί η, ε, η επιβολή θανατικών καταδικών και ισόβιων καθήρξεων σε πολλά μέλη των αδερφών μουσουλμάνων και επίσης ε, έχουν υιοθετηθεί πολλές αυθαίρετες ε, αποφάσεις από τον Ιούλιο του 2013. Εξοχότατε, Μέγα Μουφτή της Αιγύπτου, έχετε το λόγο. شكرا Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο ενώπιον των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Πολλά κράτη στον κόσμο είναι θύματα τρομοκρατίας των εξτρεμιστών, των όσων σκοτώνουν στο όνομα της θρησκείας. για το Ισλάμ θέλουμε να υπάρξει συμφιλίωση ανάμεσα στην πραγματικότητα του Ισλάμ και την πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου. Για μας κάτι τέτοιο είναι επίγουσα ανάγκη και το Πανεπιστήμιο Αλ-Ζάχαρ έχει από το 17ο αιώνα ε, εγγύψει σε αυτό το θέμα υπό την αιγίδα της εξοχότητάς του Μοχάμετ Αμπτού Αζέρ και πολλές ε, προσωπικότητες και διανοούμενοι έχουν ε, ασχοληθεί με αυτά τα θέματα στο πανεπιστήμιό μας. Πρόκειται για το θρησκευτικό ακαδημαϊκό κέντρο που είναι το παλαιότερο, διότι επισήμως αυτό λειτουργεί από το 1885. Στο πλαίσιο αυτού του κέντρου κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε ώστε να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τα ε, χάσματα ανάμεσα στην, ε, στην, στην Ισλαμική θρησκεία και τον σύγχρονο κόσμο. Εκδίδουμε φάτουα ε, όσον αφορά τις γυναίκες, τον τρόπο ντυσίματός τους. Καταδικάζουμε τη βία κατά των γυναικών. Αυτές οι Αυτά τα φάτουα έχουν δημοσιευθεί, αυτές οι, οι αποφάσεις μας και αποτελούν κομμάτι του ηθικού μας χάρτη. Επίσης έχουμε ενισχύσει τις σχέσεις και τις επαφές ανάμεσα στον χριστιανισμό και τον ε, Ιουδαϊσμό καθώς και την Ισλαμική θρησκεία αλλά και άλλες ε, ανατολικές θρησκείες. Έχουμε καταδικάσει απερίφραστα την δολοφονία αθώων κατά τη διάρκεια των 80 και του 90 και ακόμα και σήμερα συνεχίζουμε να καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή τρομοκρατίας. θέλουμε να ενισχύσουμε τις επαφές μας σε τα κοινά μας σημεία, τα όσα μας ενώνουν και να σεβαστούμε τις διαφορές ανάμεσα στις αξίες μας, αλλά Δεν μπορούμε αυτό να το καταφέρουμε παρά μόνο αν αναγνωρίσουμε αυτές τις διαφορές και τις ε, ιδιαιτερότητες που υπάρχουν ανάμεσά μας, ιδιαιτερότητες ε, που χαρακτηρίζουν κάθε χώρα, κάθε κοινωνία. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να συμβιώσουμε. Όταν ε, κανείς ε, εξετάζει αυτόν τον μεταλλασσόμενο κόσμο, τα, δει το τι συμβαίνει στη Δύση και στην Ανατολή, διαπιστώνει πως ε, τα απαραίτητα διαβήματα, τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσουν όλα αυτές η καλή θέληση να μετατραπεί σε συγκεκριμένα πράξεις ε, χρειάζεται μεγάλη ε, δύναμη για να μπορέσει, εννοείται ότι ε, για να μπορέσει το Ισλάμ να αποτελέσει έναν φορέα πρώτης τάξης που θα πρέπει οι ουλεμά, αυτοί δηλαδή που έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται στο όνομα του Ισλάμ, να μιλούν με μια φωνή. Το να ακούει κανείς τον ε, Τάδε ή τον Δίνα και να ισχυρίζεται ε, ότι αυτός εκφράζει το Ισλάμ, αυτός μιλά στο όνομα του Ισλάμ, αυτό μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση τη τόσο σοβαρή, σε αυτές τις διώξεις και τις απειλές που σοβούν σήμερα. Σίγουρα γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή, και εδώ μάλλον και κάποιο καιρό, βλέπουμε να αναδύονται διάφορα σε ομάδες όπως το, e- το ε, το οποίο μετατράπηκε σε ε, Ισλαμικό κράτος, το οποίο είναι ένας χαρακτηρισμός που μόνο του ε, έδωσε αυτό το κίνημα. Εμείς ε, δεν αναγνωρίζουμε αυτό το κίνημα. Όλα αυτά, όλες οι πράξεις του, όλες οι ενέργειές του είναι απόλυτα ε, αντίθετε με το Ισλάμ. Δεν θα πρέπει να, να, να ακούει κανείς και να εμπιστεύεται όλους όσους ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν το Ισλάμ και ότι εκφράζουν το Ισλάμ. Όλοι μας ε, είμαστε υπεύθυνοι για την κατάσταση που επικρατεί ούλεμα θα πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης του με επαγγελματισμό και ταυτόχρονα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκφράζουν την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους στο πλευρό των θρησκευόμενων, ούτω ώστε το Ισλάμ, το Ισλάμ το οποίο εκτιμάμε το Ισλάμ μας, αυτό το οποίο μας προσανατολίζει και μας καθοδηγεί, να είναι αυτό το οποίο ακούγεται. Και έτσι αυτές, αυτά τα μειονοτικά κινήματα και οι ιδέες τους να μπουν στην άκρη, να παραμεριστούν. Όλα αυτά είναι πολύ διαφοροποιημένα. Θα πρέπει πραγματικά να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να ρίξουμε τα θεμέλια μιας νέας συνεργασίας που θα περνά από πολιτιστικές, οικονομικές και ε, κοινωνικές επαφές. Χρειάζεται διάλογο σε όλους αυτούς τους τομείς ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κοινό έδαφος. Πρέπει επίσης να θεσπίσουμε ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ακαδημαϊκά κέντρα και τους φοιτητές της ε, Αιγύπτου και των άλλων χωρών, γιατί πιστεύουμε πως οι ανταλλαγές αυτές ανάμεσα στους νέους είναι εξαιρετικά σημαντικές έτσι ώστε να μην υπερισχύσει να μην υπερισχύουν οι ριζοσπαστικές αυτές θέσεις. Κάθε επαφή, κάθε συνάντηση να ε, ενισχύεται μέσω των επαφών των νέων των διαφόρων χωρών. Όταν διοργανώνουμε τέτοιου είδους συνελεύσεις των νέων, ε, διαπιστώνουμε ότι σημειώνεται μεγάλη πρόοδος κάθε φορά. Επίσης ε, θα θέλαμε να υπάρξει μια ισορροπημένη διπλωματία που θα προσεγγίσει τον Ισλαμικό κόσμο στην Δύση. Σε αυτό βασιζόμαστε πολύ γιατί ελπίζουμε πως ε, τα κράτη δικαίου, το κράτος δικαίου μάλλον, θα γίνει σεβαστό. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στη δικαιοσύνη, όποιες και αν είναι οι πεπιθήσεις μας, οι φιλοί μας, το χρώμα μας. Όλα αυτά όμως εξατμίζονται ενώπιον αυτής της σημαντικής αρχής που έχει μεγάλη αξία για μας και Κατά τη γνώμη μου νομίζω πως σε αυτά θα πρέπει να σταθώ για την ώρα και είμαι στην διάθεσή σας ε, ώστε να μπορείτε να παρέμβετε γιατί υποψιάζομαι πως θα έχετε πολλά ερωτήσεις ε, και απορίες να διατυπώσετε σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εξοχότητα για τις παρουσιάσεις σας, την παρουσίαση αυτή. Θα δώσω το λόγο στον συντονιστή από πλευρά του ΕΛΚ, τον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξοχότατε. Ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψή σας. Σημειώνουμε την έκκλησή σας προς μετριοπάθεια και ένα μετριοπαθές Ισλάμ και είναι αξιοσημείωτη και αποφασιστικότητά σας γιατί αρνηθήκατε να εγκρίνετε ε, την θανατική καταδίκη πολλών αδερφών μουσουλμάνων. Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητά σας σίγουρα, αλλά επισημαίνει και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της Αιγυπτιακής κοινωνίας. Το γεγονός δηλαδή ότι η λειτουργία της δικαιοσύνης ε, χαρακτηρίζεται από έλλειψη πιστικών αποδείξεων, πιστικών τεκμηρίων. Είναι ένα πιο γενικό πρόβλημα, ένα γενικότερο πρόβλημα της Αιγυπτιακής ε, δικαιοσύνης που πολύ πιθανόν ανακύψει και στη δίκη κατά του Μόρση. Γιατί κατηγορήθηκε για κατασκοπία λόγω συνεργασίας με τη Χαμάς και με την Ιρανική Δημοκρατία και τώρα κατηγορείται ότι πούλησε κρατικά μυστικά στο, Κατάρ. Σωρία κατηγοριών πώς τις ε, βλέπετε στο πλαίσιο του γενικότερου προβλήματος ε, της ε, απονομής της Αιγυπτιακής δικαιοσύνης. Επίσης, πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο της Τουρκίας στο μέλλον στην ευρύτερη περιοχή και σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για την επίσκεψή σας. Ο κύριος Καν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την παρουσία σας εξοχότατε. Έχω δύο ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Ακούσαμε για την Αραβική Άνοιξη και είδαμε τις αλλαγές που γίνονται και την κατάσταση στην Αίγυπτο που έχει πολύ σημαντική θέση στον αραβικό κόσμο. Πιστεύετε ότι παρατηρείτε μία παλιδρόμηση και πώς πιστεύετε ότι μπορούν να έχουν περισσότερο λόγο οι πολίτες ε, για τους κυβερνώντες τους. Μιλήσατε για το ίσις, για το Ισλαμικό κράτος. Είναι σαφές ότι η ρητορική που χρησιμοποιεί το Ισλαμικό κράτος είναι θρησκευτικού χαρακτήρα. Το ύφος τους είναι θρησκευτικό. Οι δράσεις τους όμως αντιβαίνουν στις θρησκευτικές αξίες που επικαλείται το Ισλαμικό κράτος και πολλοί νέοι, όχι μόνο από το Ισλαμικό κόσμο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζονται από την ε, ρητορική αυτή. Πώς, πώς μπορούν να δράσουν ε, και το Πανεπιστήμιο Αλζαχάρ και άλλα μουσουλμανικά Ινστιτούτα, ώστε να φτάσει στους νέους το πραγματικό μήνυμα του Ισλάμ και όχι αυτό το μήνυμα το ψεύτικο του Ισλάμ που δίνει το Ισλαμικό κράτος. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και εδώ είμαι η εξοχότητά σας και φυσικά συμφωνώ με όσους ε, ανακοίνωσαν και είπαν την θαυμασμό τους σε ό,τι αφορά τους Σουνίτες του Σουλέμα. Και το θέμα αυτό με απασχολεί επί σειρά ετών σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, την ανεκτικότητα, σε ό,τι αφορά την τάγματα των όντων για την επιβολή θεματικών θεματικής ποινής μετά από βλασφημία, μετά από απιστία, μοιχεία και δυστυχώς αυτό συχνά επιβάλλεται σε μειονότητες, ιδιαίτερα στους χριστιανούς. Πώς μπορεί λοιπόν το δόγμα του Ιστιχάτ ε, να επιτρέψει, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Φυσικά υπάρχει το θέμα της αντικής ποινής ε, μεταξύ πολλών Ισλαμικών χωρών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμβιβαστούμε σε κάποιο με κάποιο τρόπο προκειμένου να καταργηθεί αυτή η εξαιρετικά σκληρή ποινή για όσους δεν θέλουν να έχουν θρησκεία ή θέλουν να αλλάξουν την θρησκεία τους σε ό,τι αφορά το θέμα του Ισλαμικού κράτους, ε, του ISIS, ε, που είναι πολύ σημαντικό για μας ε, στη χώρα μου, στο Βελγίο, στη Γαλλία, γιατί είναι χιλιάδες Βρετανοί που αγωνίζονται υπέρ της ίσας και Πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα ε, εξεδόθη η ΦΕΤΒΑΣ προκειμένου να είναι απαγορευμένη η προσχώρηση των Βρετανών πολιτών στον, στην οργάνωση αυτή. Θα ήσασταν ιτεθειμένος να επαναλάβατε την ε, καταδίκη τέτοιων τρομοκρατικών ε, κινημάτων και να α, καταδικάσατε τον κ. Μπαγκάτη ως αυτόν κ. Χαλίφη, δεδομένης της κατάστασης. Γιατί και αυτός και η οπαδή του επιβάλλουν ένα μεσονικό καθεστώς, τρόμο κατά των ε, χριστιανών, των των ε, μουσουλμάνων, του γιαζίτη, των ε, Αρμενιών, των Εβραίων και το καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το πάρα πολύ τρομακτικό και αυτό φυσικά αποτυπώνεται και σε ό,τι αφορά την περιφερειακή αλλά και την παγκόσμια ασφάλεια. Desde hace decenios. Εδώ και δεκαετίες ε, γινόμαστε μάρτυρες μιας ομογενοποίησης ε, ε, πολιτιστικής και θρησκευτικής του αραβικού κόσμου. Έχει χαθεί τεράστια συνεισφορά της εβραϊκής κοινότητας. Χάνεται η χριστιανική παρουσία, δημιουργείται, δημιουργούνται κάποιες κοινότητες που εγκλωβίζονται στον εαυτό τους και οι Σίτες και οι Σουνίτες μεταξύ τους αισθάνονται εχθρότητα σε πολλά μέρη και εχθρότητα και κατά των Δρούζων και των, των Αλαβητών. Και χωρίς τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι αδύνατο να αντιληφθούμε την εξέλιξη της, του αραβικού πολιτισμού αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού. Και μάλιστα το Αιγυπτιακό Κομμουνιστικό Κόμμα ιδρύθηκε από έναν Εβραίο της Αλεξάνδρειας αυτή τη στιγμή χάνονται όμως κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής και κοινωνικής συνεισφοράς. Ε, γιατί χάνουμε τους συνεστόριους στο Ιράκ, τους χριστιανούς που είναι πια μειονότητα στην Βιθλέμ και τους ε, και χριστιανούς που φεύγουν από την Παλαιστίνη είναι δύσκολο να καταλάβουμε τον αραβικό κόσμο χωρίς την πολυμορφία, τη θρησκευτική και την εθνοτική. Όταν η Ισπανία έδιωξε τους σεφαρδίτες ε, Εβραίους, ε, ο Ισλαμικός και ο αραβικός κόσμος άνοιξαν τις αγκάλες τους. Επίσης, τι εναλλακτικές λύσεις έχουν οι κόπτοι της Αιγύπτου που αντιμετωπίζουν δυσκολίε σε πολλές ζώνες τη Αιγύπτου και στο ίδιο το Κάιρο μερικές φορές. Είναι πραγματικά τραγική και θλιβερή αυτή η κατάσταση διάσπασης που υπάρχει στην αραβική κοινωνία και ε, εξάλληψης μερικών σημαντικών κοινοτήτων, ειδικά από κάποιες αυτοαποκαλούμενες ομάδες προστασίας. Θα ήθελα επαναλάβω την χαρά μου για την παρουσία του του και θα ήθελα να πω ότι πρόσφατα εγκρίναμε ένα καταπήγον ψήφισμα ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την προστασία των ε, ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ε, καταδίκη, επισημάνεται την καταδίκη δημοσιογράφων και τη σύλληψή τους και το θέμα της θανατικής ποινής. Ε, τι γνώμη έχετε για αυτή τη, τη δημοκρατική παρεκτροπή που διαπιστώνω αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο. Επίσης, τι γίνεται με την επιρροή στις υπόλοιπες αραβικές χώρες. Πώς πιστεύετε θα πρέπει να οργανωθούν οι αραβικές χώρες για να αποφύγουν τους θρησκευτικού αγώνες. Έχετε ένα μοντέλο κατά νου ή είστε σε θέση να προτείνετε ένα μοντέλο για να αποφευχθούν τέτοιες θρησκευτικέ διαμάχες. Ε, Your Excellency ε, Εξοχότητά σας, ε, μεγάλη μουφτή της Αιγύπτου. Θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση για τη δημοκρατία. Είσαστε ο πρώτος δημοκρατικά αιρετός μεγάλος μουφτής της Αιγύπτου. Και το ίδιο ισχύει για όλους τους ευρωβουλευτές που βρίσκονται εδώ πέρα στην αίθουσα. Κάποια τμήματα της ελλαμικής κοινωνίας διατείνονται ότι η δημοκρατία δεν έχει ρόλο στο Ισλάμ και προτείνουν άλλες ε, λύσεις. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας γνώμη για τη δημοκρατία. Κατά δεύτερον, ποιος θα είναι ο ρόλος σας κατά τα δέκα χρόνια που θα διτελέσετε μεγάλο μουφτή τη Αιγύπτου. Τι κληροδότημα θέλετε να αφήσετε πίσω σα. Και κατά τρίτον, θα ήθελα να σα καλέσω ω φωνή τη ε, μετριοπάθεια σε μία σύνοδο στο Λονδίνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλέσετε την νεολαία που ριζοσπαστικοποιείται με τη φωνή της μετριοπάθειας να ακολουθήσει αυτή την ε, οδό. Και θα ήθελα να σας καλέσω να είστε κύριος ομιλητής αυτή την, ε, σε αυτό το συνέδριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξοχότατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ σημαντικά σας λόγια που έχουν ε, ιδιαίτερο νόημα σε αυτό το σώμα από πλευράς ενός βουλευτή που πιστεύει στα όσα μας δίδαξε ο για τη σημασία μιας βασικής ε, έννοιας της ε, οριζόντιας ενότητας των ε, θρησκειών. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη όπως ε, εξάλλου πιστεύω αυτό υπονοείται και στην θέση που λάβατε, σκοπεύετε πέρα από μια θεωρητική καταδίκη, θα κάνετε και μια πιο δραστήρια δράση όσον αφορά την υπεράσπιση των χριστιανών που διώκονται σε πολλές περιοχές του αραβικού ισλαμικού κόσμου. Δεύτερο πιο συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά την κατάσταση που θα έλεγα προηγείται της στρατολόγησης εξτρεμιστών τρομοκρατών μέσω οργανώσεων ε, του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το, το κήρυγμα από πλευράς πολλών, πολλών πολυάριθμων σε διάφορα μέρη και διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, ε, ε, δηλαδή κηρυγμάτων που κάνουν διάφοροι ημάμας, ημάμιδες που από μόνοι τους έχουν αυτά να κηρυχθεί ως εκπρόσωποι του Ισλάμα, μεταξύ αυτών και στη χώρα μου στην Ιταλία, αυτοί κάνουν μια διαρκή προπαγανδιστική δράση εξτρεμιστική που χρησιμοποιεί, χειραγωγεί την ε, ορολογία και φυσικά στρεβλώνοντας ε, τα διδάγματα του Κορανίου με στόχο να ε, μπορέσουν να στρατολογήσουν τους νέους για τρομοκρατικές ενέργειες. Πιστεύω πως είναι απαραίτητη και επίγουσα μια συγκεκριμένη δράση όχι μόνο μέσω της διδαχής και των προσανατολισμών και των ενδείξεων που προέρχονται από τις επίσημες πηγές του Ισλάμ, αλλά πάντως συγκεκριμένη δράση ώστε να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτού του είδους τη δραστηριότητα και την ε, ε, ε, ελεύθερη ε, κυκλοφορία αυτών των ε, ε, αυτό, ανακηρυσσόμενων εκπροσώπων του Ισλάμ. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι συντονισμός και δράση έτσι συγκεκριμένη και κέρια για κατευθύνσεις ε, προς την ε, εξάλληψη ενός τόσο σημαντικού κινδύνου, ε, μια στρέβλωση η οποία είναι δυσφημιστική προς το αληθινό Ισλάμ. Μια τέτοια δράση λοιπόν δεν έχει γίνει ακόμα. Ο κύριος Πέτερλε. Εξοχότατε. με χαροποίησε το γεγονός ότι σταθήκατε ιδιαίτερα στην ανάγκη του διαλόγου. Είμαι μέλος του φόρουμ που έχει η ομάδα μου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για το θρησκευτικό διάλογο. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να εμβαθύνουμε αυτό το διάλογο, αν θέλουμε ε, να βελτιωθεί η κατάσταση. Είχα πάει στην Ιγυρία και την Κένια σε αποστολές παρατήρηση εκλογών και είχα συνομιλίες με μουσουλμάνους που εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάκριση εξουσιών και για τη διαχωρισμό του κράτους από τη θρησκεία. Με ενδιαφέρει λοιπόν ποιος είναι ο συνομιλητής μας για τα θέματα αυτά, γιατί μερικοί δεν επιθυμούν το διάλογο, προτιμούν τη βία αντί για το διάλογο. Εσείς ποιος πιστεύετε θα πρέπει να είναι ο συνομιλητής μας, ο συνομιλητής Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή για τα θέματα αυτά. Μάλιστα, Πρόεδρε. Μεγάλε ε, μουφτή, ε, βρίσκομαι εδώ. Να, εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε μέχρι εδώ και να σας πω, όπως είπε προηγουμένως και ένα συνάδελφος, πως είναι αλήθεια ότι είναι σημαντικό να είστε ο πρώτος μεγάλος μουφτής που δεν έχει διοριστεί από τον πρόεδρο, αλλά που εξελέγει από το, Συμβούλιο, το Ισλαμικό Συμβούλιο Ακαδημαϊκών. Και πάλι θεωρώ δηλαδή ότι εδώ ε, σας αποδίδεται μια νομιμότητα που είναι θεμελιώδη σημασία. Θα ήθελα να σας υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Ε, χαιρετήσατε και χαιρετίζω και εγώ την σαφή σας καταδίκη του Ισλαμικού κράτους. Είναι σημαντικό μια θρησκευτική προσωπικότητα όπως εσείς να βρει τα σωστά λόγια ώστε να καταδικάσει αυτή την απειλή. Διαπιστώνουμε ότι οι Αιγυπτιακές ε, ομάδες έχουν ήδη δηλώσει σύμμαχοι του Χαλίφη Ουμπραήμ όπως η Παρτιζάν της Ιερουσαλήμ που είναι εγκατεστημένη στο Σινά. Θέλω να γνωρίζω ποιος, ποιος είναι ο αντίκτυπος όλων αυτών για την ε, Αίγυπτο. Δεύτερη ερώτηση. Είστε αντίθετος στη θενατική καταδίκη πολλών εκατοντάδων ε, αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο. Ήταν μια θεραλέα αλλά απαραίτητη απόφαση. Βλέπετε να υπάρχει κάποια ε, ηρεμία στην κοινωνία την Αιγυπτιακή και πώς το Ευρωπαϊκό μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή τη ε, διαδικασία ειρήνευσης Έπειτα, ε, κάποιοι εξομοιώνουν το σύνολο των αδερφών μουσουλμάνων με τους τρομοκράτες. Εσείς πριν από λίγο μιλήσατε για τον ε, ηθικό χάρτη, για την καταδίκη κάθε είδους τρομοκρατή. Εσείς ελπίζετε πως θα υπάρξει μια αύληνση των καταδικών κατά των αδερφών ε, μουσουλμάνων, ιδιαίτερα μετά τη δήλωσή σας. Σας χαιρετίζω ε, εξοχότατε και πολύ θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις που θα δώσετε στους συναδέλφους ε, όσον αφορά την καταστολή και την φυλάκιση των δημοσιογράφων. Το ερώτημά μου είναι για τις γυναίκες. Είπατε πως η προσπάθειά σας είναι να συμφιλειωθεί η θρησκεία με τον σύγχρονο κόσμο και ο σύγχρονος κόσμος αναγνωρίζει τις γυναίκες βεβαίως ως απόλυτες δικαιούχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλες ελπίδες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες στην Αίγυπτο που ηγούνται του κινήματος ε, για ε, της ε, πλατείας Ταχρήρ και βέβαια Υπήρξε αρνητικό αντίκτυπο. Ήμουν ε, παρόν ε, το 2011 με τον προκράτοχό σα που δεν είχε εκλεγεί, αλλά πρέπει να σα πω πω δεν ήμουν καθόλου ήσυχη όσον τι γυναίκε, όταν α πούμε διαμαρτυρηθήκαμε ότι οι γυναίκε ε, υπόκειτο σε τεστ κολπικά κτλ. Πώς βλέπετε λοιπόν την εξέλιξη των σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες στην Αίγυπτο και αλλού. Έπειτα για τη Λιβύη φυσικά τα όσα συμβαίνουν εκεί επηρεάζονται από τα όσα συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Πώς βλέπετε την κατάσταση και το κίνδυνο όταν εσείς δεν έχετε κράτος, λέει ο κόσμος για καταραίων ε, κράτος στην Λιβύη ε, και βέβαια υπάρχει μια ακόμα επικράτεια η οποία είναι ε, έρμεο της κατάχρησης από διάφορους ριζοσπαστικού ριζοσπαστικέ ομάδες και βέβαια ποιος είναι, επηρεάζεται και ο, η διάθεση των ανθρώπων και ο, ο τρόπος που ασκούν τις διαταχές του Ισλάμ. Και έπειτα, ο ρόλος των ε, θρησκευόμενων, πού είναι αυτοί, πού βρίσκονται, γιατί δεν λένε στους νέους του, του Ισλαμικού κόσμου πως όλα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν το Ισλάμ και ότι όλα αυτά είναι τελείως αντίθετα με το Ισλάμ. Σας ευχαριστώ εξοχότατε για την παρουσία σα, και για το, το ότι μας παρουσιάσατε τη θέση σα και τις απόψεις σας. Πώς κρίνετε την κατάσταση των χριστιανών στην Αίγυπτο του σήμερα και πέρυσι είχαμε πολλά θύματα βιασμών και βιοπραγιών στη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης. Ω λόγιος ε, είστε και εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά ούτε ε, η, η κοινωνία της Αιγυπτού, ούτε το Αιγυπτιακό κράτος εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει ειρήνη με το Ισραήλ. Πώς ε, παρουσιάζεται την κατάσταση αυτή και πώς διάκειται η, η Αιγυπτιακή κοινωνία απέναντι στην κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ah, danke. Εξοχότατε και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ σήμερα για το γεγονός ε, ότι μιλήσατε έτσι εισαγωγικώς με λόγια τα οποία με άκηξαν ιδιαίτερως και θα σας ευχαριστήσω που απαντάτε και στις ερωτήσεις μας. Θα φαντάζεστε ότι όλοι εδώ ανησυχούμε ιδιαίτερως ε, σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση στην Αίγυπτο. Και ως εκ τούτου λοιπόν η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξή. Ευτυχώς ε, εσείς ε, έχετε ταχθεί κατά της θανατικής ποινής που επιβλήθηκε στους αδελφούς μουσουλμάνους και σε ό,τι αφορά Άλλε ε, καθεξής. Πρακτικά, πώς θεωρείτε ότι μπορείτε και κατά πόσο είναι δυνατόν να αποτραπεί η εφαρμογή της θανατικής αυτής ποινής. Δεύτερη ερώτηση. Ακούσαμε διάφορες παρατηρήσεις εδώ σε ό,τι αφορά τους κόπτες στην Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το θέμα με τους κόπτες, αυτό το θέμα εδώ και αιώνες ε, συνεχίζεται. Πώς πιστεύετε ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση. Θα είναι δυνατόν επιτέλους να υπάρξει ειρήνευση μεταξύ των ομάδων αυτών. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι συστήνετε, τι μας συστήνετε να κάνουμε κατά της τρομοκρατίας, κατά του γεγονότος ότι όλο και πιο πολλοί νέοι από τις χώρες μας εντάσσονται στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε συμβουλές. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξοχότατε. Σαλάμα Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μας να μπορούμε να σας συναντήσουμε σήμερα και θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου εκτίμηση για το μήνυμά σας που δείχνει άνοιγμα και ελπίδα. Ε, θέλουμε όντως να υπάρξει μια κοινωνική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Χρειάζεται κατά τη γνώμη μου μια ισχυρή και δημοκρατική Αίγυπτος για να μπορέσει να αντιμετωπίσουμε τις, τοπικές, τις περιφερειακές κρίσεις που ε, θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Χωρίς μια ισχυρή Αίγυπτο δεν μπορούμε να πετύχουμε σταθερότητα και βλέπω θετικά και ένα ειρηνικό μήνυμα το οποίο καταδικάζει τις ε, μονομερείς στρατιωτικέ ε, επεμβάσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο σκοπεύετε να στηρίξετε αυτό το μήνυμα, το ειρηνευτικό, το σεβασμό για τις μειονότητες σε ολόκληρο τον Ισλαμικό κόσμο και όχι μόνο στις Ισλαμικές χώρες αλλά και στις Ισλαμικές κοινότητες που ζουν στην Δύση και σε άλλες ε, περιοχές του κόσμου. Κατά τη γνώμη σας, τι βάρος μπορεί να, έχουν, έχει η χρήση των μεγάλων μέσων ε, μαζικής επικοινωνίας, δεδομένου του κύρους ε, του λόγου σας και της προσωπικότητάς σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Ερωτήσεις που δείχνουν το ενδιαφέρον σας για την ε, θέση της Αιγύπτου αλλά και τις απόψεις ε, του μουφτή της Αιγύπτου για τα θέματα αυτά. Πρόκειται για θέματα που δημιουργούν μεγάλο προβληματισμό. Οι περισσότερες ερωτήσεις στράφηκαν γύρω από ε, το θέμα των θανατικών καταδικών ε, και τη θέση της γυναίκας, το θέμα του διαθρησκευτικού διαλόγου και το ζήτημα του Ισλαμικού κράτους. Σε ό,τι αφορά την εσχάτη των ποινών και το ρόλο του μουφτή σε σχέση με τις θανατικές ποινές. κώδικας ποινικής δικονομίας στην Αίγυπτο προβλέπει μία σειρά διαδικασιών που προστατεύει και τα, τη δικαιοσύνη αλλά και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Μπορεί να σας εκπλήσει κάτι τέτοιο, αλλά οι διαδικασίες αυτές είναι περίπλοκες και ακριβώς εξαιτία τη περιπλοκότητα της οικονομία είναι σχεδόν αδύνατο να καταλήξει κανεί σε θανατική ποινή. Θα σας εξηγήσω εν ολίγη σε αυτή τη διαδικασία. Η αστυνομία ε, αυτεπάγγελτα ενεργεί ε, ε, ενεργή και παραπέμπει το θέμα στην, στον εισαγγελέα που συντάσσει το κατηγορητήριο και η δικογραφία μεταφέρεται στο δικαστήριο. Και μάλιστα από το 1950 έχουμε και ανακριτή στην ε, διαδικασία αυτή. Οπότε ο αρμόδιος εγγελέας που ασχολείται με την ε, έρευνα και την ανακριτική διαδικασία ενεργεί το πρώτο, την πρώτη φάση της ανακριτικής διαδικασίας και στη συνέχεια το θέμα παραπέμπεται σε ένα δικαστικό συμβούλιο. Οι δικαστές είναι τρεις και αποφασίζουν για την κατάλληλη ποινή που θα πρέπει να απαγγελθεί. Πριν αποφαθούν, οφείλουν να παραπέμψουν τη δικογραφία στο μουφτή. Ο μουφτής λοιπόν λαμβάνει το σύνολο της δικογραφίας από την έναρξη της ε, διαδικασίας, την ανάκριση και την πρόταση της θανατικής ποινής από το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο μουφτής εξετάζει λεπτομεριακά όλα τα στοιχεία, το σύνολο της δικογραφίας και δίνει τη νομική του γνωμοδότηση. Η γνώμη του μουφτή δεν αφορά ούτε την ουσία, ούτε τον τύπο, ούτε τη διαδικασία. Ούτε κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, ούτε κατά τη διάρκεια της δικαστικής απόφασης. Ο μουφτής αποφαίνεται το κατά πόσο η προτινόμενη ποινή συνάδει με το Ισλαμικό δίκαιο. και δεν είναι κανείς υπέρ ή κατά της ε, θανατικής καταδίκης χωρίς να έχει αδιάστα στοιχεία, ατράνταχτες αποδείξεις. Στη συνέχεια ο Μουφτής ε, στέλνει τη νομική του γνωμοδότηση στους δικαστές που ήταν αρμόδιοι επί της ουσίας. Από τη στιγμή που το δικαστικό αυτό συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση, τη γνωμοδότηση του Μουφτή, είναι ελεύθερο να οριστικοποιήσει την γνώμη του και να λάβει υπόψη ή όχι την γνωμοδότηση του μουφτή. Οι τρεις λοιπόν δικαστές που είναι αρμόδιοι για την ουσία της υπόθεσης μπορούν είτε να δεχτούν την νομική γνωμοδότηση του μουφτή είτε να την απορρίψουν. Αλλά σε τελική ανάλυση και επί της ουσίας αρμόδιοι είναι οι δικαστές για την οριστική απόφαση. Οι δικαστές επιδικάζουν την ποινή ή όχι. Λαμβάνοντας ή όχι την νομική γνωμοδότηση του μουφτή. Αλλά σε τελική ανάλυση ο δικαστής κρίνει. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντιφατικές ποινές υπάρχει δυνατότητα έφεσης. Ακόμη και ο εισαγγελέας αυτεπάγγελτα μπορεί να υποβάλει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο. που είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο στην Αίγυπτο. Και μάλιστα περίπου 99% των δικαστικών αποφάσεων ακυρώνονται. Και παραπέμπονται σε άλλο ποινικό δικαστήριο. Και μάλιστα μετά την ακύρωση της διαδικασίας γίνεται επανεξέταση και της ουσίας της υπόθεσης. Αν το νέο ποινικό δικαστήριο θεωρεί και πάλι ότι επιβάλλεται να επιβληθεί θανατική ποινή, θα πρέπει και πάλι να στείλει το σύνολο της δικογραφίας στο μουφτή. Ο μουφτής εξετάζει εκ νέου όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και εκδίδει μια δεύτερη δικαστική, νομική συγγνώμη, γνωμοδότηση, την οποία στη συνέχεια στέλνει στο δεύτερο αυτό ποινικό δικαστήριο. Αν και τη δεύτερη φορά ο δικαστής επικρίνει, ε, επικυρώσει την πρώτη θανατική καταδίκη, ε, το θέμα παραπέμπεται και στον πρόεδρο της ε, Δημοκρατίας που πρέπει και αυτός να κυρώσει τη θανατική ποινή. Η όλη διαδικασία διαρκεί μια τετραετία. Χρειάζεται μια τέτοια χρονοβόρα διαδικασία σε περίπτωση που επιβάλλεται μια τόσο σοβαρή ποινή όπως είναι η θανατική. Στατιστικά λοιπόν, σε ελάχιστες περιπτώσεις εκτελείται μια τέτοια θανατική καταδίκη. Και εδώ μιλούμε για ε, διαδικασίες που, υπήρχε, που γινόταν κατά αντιμόλια. Αν τώρα έχουμε έρημο δικίες και αν στη συνέχεια συλληφθεί ο κατηγορούμενος, θα πρέπει να ξαναρχίσει εκ νέου διαδικασία. Ακόμη και αν έχει εκδοθεί απόφαση ερήμην αρχικά του κατηγορουμένου. Φυσικά όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Και μερικές φορές το διαπραχθένα έγκλημα δημιουργεί μια κατάσταση, ένα κλίμα τρόμου και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και φυσικά θα πρέπει να δείχνουμε ευσπλαχνία και έλεος, αλλά τη στιγμή που κρίνουμε ένα έγκλημα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θύμα. Το θύμα που ενδέχεται να έχασε τη ζωή του, που στερήθηκε το δικαίωμα της ζωής. Ενδεχομένως το θύμα είχε οικογένεια, είχε παιδιά. και έχασε την ευκαιρία αυτή να συνεχίσει τη ζωή του. Όταν λοιπόν εξετάζουμε όλες αυτές τις περιστάσεις, έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, τότε διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται και η θανατική ποινή. Και πολλοί Ευρωπαίοι φιλόσοφοι σε πραγματείες τους μίλησαν για την φιλοσοφία του εγκλήματος και τη φιλοσοφία της ποινή. Και το Ισλάμ υιοθετεί αυτή τη φιλοσοφία της ποινή. Θεωρούμε ότι η θανατική ποινή έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα. Και φυσικά όταν κάποιος ε, στερεί τη ζωή σε κάποιον άλλον, μερικές φορές ε, αξίζει και θανατική ποινής. Αυτά ως προς την ε, ποινική διαδικασία. Τώρα, επί του παρόντος, η Αίγυπτος, σας μιλάω ειλικρινά, διανύει μια αρκετά σταθερή περίοδο. Μάλιστα είχαμε δύο σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν το Σύνταγμα. Είχαμε καταρχήν τη, τη σύνταξη του Αιγυπτιακού Συντάγματος και τη λαϊκή ετοιμιγορία για το Σύνταγμα του 2014. Μάλιστα και εγώ προσωπικά συμμετείχα στη σύνταξη του νέου συντάγματος. Συμμετείχα στην ε, γνωστή ομάδα των 50 και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ήταν πολύ θετικά και έδειξαν την έγκριση του Αιγυπτιακού λαού για το Σύνταγμα. Η δεύτερη σημαντική ημερομηνία ήταν η ημερομηνία των προεδρικών εκλογών. Και από αυτού θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των κοπτών στην Αίγυπτο, στο θέμα της κοπτικής κοινότητας. Επαναλαμβάνω, κάθε υπήκος της Αιγύπτου είναι πρώτα απ' όλα Αιγύπτιος επίκος. Δεν έχουμε την έννοια των μειονοτήτων και περισσότερο λαμβάνουμε υπόψη την εθνότητα παρά την θρησκευτική συμμετοχή σε κάποια θρησκευτική κοινότητα. Ο πολιτισμός μας είναι ανοιχτός προς όλες τις θρησκείες. Αυτό έχει δείξει και η ιστορία μας. Και η ιστορία προϋποθέτει μία πολυμορφία. Δεν μπορεί κανείς να γεμίσει την ιστορία μόνος του. Χρειαζόμαστε όλους τους φορείς της Αιγυπτιακής κοινωνίας. Έτσι διαμορφώνουμε την ιστορία μας. Γιατί στην Αίγυπτο συνυπάρχουμε και μάλιστα σχεδόν ιδεοδός συνυπάρχουμε στις συνοικίες μας, στα πανεπιστήμια μας, στα σχολεία μας και δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Δεν κάνουμε διακρίση με αυτούς τους όρους, ούτε στο χώρο της εκπαίδευσης, ούτε στο χώρο της εργασίας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Δεν ξέρουμε ποιος είναι χριστιανός και ποιος είναι μουσουλμάνος. Θα ήθελα να σας Καθησυχάσω λοιπόν ότι η κοπτική κοινότητα αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της Αιγυπτιακής κοινωνίας και του Αιγυπτιακού πεπρωμένου και είμαι ένθερμος υποστηρικτής του κράτους δικαίου. Πιστεύω ότι αυτή η αρχή του κράτους δικαίου θα πρέπει να πριτανεύσει και όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά παντού. Ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς καμία διάκριση. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση των γυναικών στην Αίγυπτο. Έχω δημοσιεύσει πολλές έρευνες για το θέμα αυτό, την κατάσταση των γυναικών στην Αίγυπτο και τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών στην Αίγυπτο, καθώς και τα δικαιώματα των γυναικών στο γάμο. Οι γυναίκες απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματα που απορρέουν ε, από την ιδιότητά τους ως πολίτη και ως ε, συζύγου. Και μάλιστα ο προφήτης Μωάμε θα αναφέρεται στις γυναίκες ως συντρόφους των ανδρών. Και το Κοράνι δεν διαχωρίζει τους άνδρες από τις γυναίκες. Απευθύνεται και στους δύο. Φυσικά υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Κάποιες θρησκευτικές πρακτικές απαγορεύονται για τις γυναίκες σε συγκεκριμένες περιόδους. Υπάρχουν περίοδοι που η γυναίκα δεν μπορεί ούτε να νηστέψει ούτε να προσευχηθεί. σε ό,τι αφορά την Ισλαμική νομολογία, και τον Ισλαμικό νόμο υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και το Αιγυπτιακό Σύνταγμα το 2014 επέμεινε ιδιαίτερο στο σημείο αυτό της ισότητας. Μάλιστα υπάρχει και ειδικό άρθρο, ιδιαίτερα λεπτομεριακό, για να αποφεύγονται παρερμηνίες στην Αιγυπτιακή νομοθεσία και να μην παραβιαστούν τα δικαιώματα των γυναικών ή να μην επιδεινωθεί η θέση των γυναικών. Επαναλαμβάνω, οι γυναίκες απολαμβάνουν ε, πλήρως τα δικαιώματά τους και ίσως σε λίγα χρόνια οι άνδρες θα διεκδικήσουν κάποια δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ίσις, η Ισλαμικό κράτος και τις δραστηριότητες ε, του Ισλαμικού κράτους και του αυτοποκαλούμενου Χαλίφη Αλμπαγδάδη. Θα προτιμούσα να μην μιλήσω καν για χαλιφάτο, ούτε να αναφερθώ σε κράτος, Ισλαμικό κράτος. Γιατί δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που να στοιχειοθετούν την ύπαρξη ενός κράτους. Και αναλύοντας τις δράσεις αυτής της οργάνωσης που αποκαλείται Ισλαμικό κράτος, αν αναλύσουμε επιστημονικά αυτές τις δράσεις, και υπό το φως ε, των αρχών και των αξιών της Ισλαμικής θρησκείας διαπιστώνουμε ότι οι δράσεις αυτής της οργάνωσης συνιστούν αξιόπινες ενέργειες, εγκληματικές ενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμος και με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου να διωχθούν αυτοί οι άνθρωποι, τα μέλη αυτής της οργάνωσης και να δικαστούν ανάλογα με την σοβαρότητα των πράξεών τους. Δεν υπάρχει κανένα θρησκευτικό κείμενο στο Ισλάμ που ε, να εξυμνάται η δράση, η βία, η καταστροφή ή να γίνεται παρότρινση για δολοφονία ή άσκηση βίας. Κανένα θρησκευτικό κείμενο δεν περιλαμβάνει τέτοιες παρενέσεις. Το Ισλάμ ε, μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου από έναν άντρα και μία γυναίκα. Και οι πιο ευγενείς άνθρωποι είναι και οι πιο ευσεβείς άνθρωποι. Ο Θεός θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει μία μόνο κοινότητα, μία μόνο θρησκευτική κοινότητα, μία μόνο ε, πίστη. Αλλά επέτρεψε ακριβώς αυτή την θρησκευτική πολυμορφία. Γι' αυτό και εμείς ε, εξασφαλίζουμε την ανεξιθρησκεία. Και στο Σύνταγμά μας υπάρχει ένα άρθρο που αποτέλεσε τον καρπό μακροχρόνια συζήτησης και που εξασφαλίζει την ανεξιθρησκεία και την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει στη θρησκεία του αλλά οι δράσεις του θα πρέπει να εντάσσονται στο κράτος δικαίου. Οπότε οι δράσεις της Ισλαμικής αυτής οργάνωσης που αποκαλείται Ισλαμικό κράτος δεν δικαιολογούνται με βάση τις αρχές του Ισλάμ. Πρόκειται για μία οργάνωση που καπηλεύεται τη θρησκεία, την Ισλαμική θρησκεία. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα θρησκευτικό κείμενο του Ισλάμ που να ε, ζητά απελάσεις πληθυσμών ε, διώξεις κοινοτήτων ή οτιδήποτε τέτοιο. Και μάλιστα ακόμη και σε περίοδους πολέμου επιτρέπεται η δίωξη μόνο των μαχητών. Και μάλιστα οι γυναίκες δεν εντάσσονται στο μάχημα πληθυσμό, είναι άμαχος πληθυσμός. Το Ισλάμ απαγορεύει της διώξεις αμάχου πληθυσμού ή τη δολοφονία αμάχου πληθυσμού. Ή ιερέων που βρίσκονται σε θρησκευτικούς χώρους. Απαγορεύεται η τη δολοφονια αμαχου πληθυσμου οι ιερεων που βρισκονται σε θρησκευτικους χωρους απαγορευεται η επιθεση στον άμαχο πληθυσμό, απαγορεύεται ακόμη και η κατεδάφιση ενός σπιτιού ή το κόψιμο ενός δέντρου. Μπορώ να σας παραπέμψω σε θρησκευτικά κείμενα του Ισλάμ που περιλαμβάνουν όλους αυτούς τους περιορισμούς και που δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη και στον πόλεμο μια συγκεκριμένη ηθική που θα πρέπει να τηρείται. Ακόμη και σε εμπόλεμες καταστάσεις, ακόμη και σε ένοπλες ε, σειράξεις ή στο, εσωτερικό μιας χώρας ή μεταξύ διαφόρων χωρών, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες ηθικές αρχές. Οι πράξεις της ε, οργάνωση Ισλαμικό κράτος σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τις αρχές του Ισλαμ, του Ισλάμ και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από το Ισλάμ. Σε ό,τι αφορά την μαζική αποχώρηση χριστιανών από την Αίγυπτο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένο φαινόμενο. μπορεί να υπάρχει κάποια πίεση, αλλά όπως σας είπα υπάρχει πολύ ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. Για παράδειγμα, ο δόκτωρ Ναμπί Λόκα είναι χριστιανός. Διαβάζοντας το βιογραφικό αυτής της ιστορικής προσωπικότητας, διαπιστώνουμε ότι ως παιδί πήγαινε σε Ισλαμικό σχολείο, ενώ ήταν χριστιανός. Είναι χριστιανός. Έγραψε όμως βιβλίο για τη ζωή του Μωάμεθ με τίτλο «Μωάμεθ, ο προφήτης και το μήνυμα». Εκεί παρουσίασε τις θετικές πτυχές του Ισλάμ, παρόλο που ήταν χριστιανός και έμεινε χριστιανός μέχρι το θάνατό του. Πολλοί ηγέτες του Ισλαμικού κόσμου σε κά... γεννήθηκαν από μητέρες που ήταν χριστιανές. Κάτι που δείχνει τις σημαντικές αλληλεπιδράσεις, τις βαθύτερες αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στην Αιγυπτιακή κοινωνία σεβόμαστε πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και, τα δι... και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Για παράδειγμα, το Αιγυπτιακό Σύνταγμα του 2014 έχει ειδικό κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για πρώτη φορά στην ιστορία μας και μπορεί να σας εκπλήσει αυτό το γεγονός γιατί γνωρίζω ότι οι διεθνείς συνθήκες λαμβάνουν υπόψη, λαμβάνονται υπόψη στις εθνικές ένομες τάξεις. Εμείς λοιπόν αναφερθήκαμε στην ανάγκη να τηρήσουμε τα άρθρα των διεθνών συνθήκων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και Δεσμευθήκαμε να τηρήσουμε όλες τις διεθνείς συνθήκες που υπέγραψε η Αίγυπτος. Γιατί το Κοράνιο μας ενθαρρύνει και μας επιβάλλει την τήρηση των συμφωνιών που έχουμε αναλάβει. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας. Και ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος, η αλλαγή της κυβέρνησης στην Αίγυπτο, τηρήθηκε η ειρηνευτική συμφωνία που είχαμε συνάψει με το Ισραήλ, άσχετα με την ε, αλλαγή στις κυβερνήσεις. Η δημοκρατία είναι ένας ε, σύγχρονος μηχανισμός για τη διαχείριση της εξουσίας. Εμείς προσπαθούμε με την προσέγγισή μας να διαπιστώσουμε κατά πόσο η δημοκρατία επιτρέπει στην κοινωνία να απολαύσει κάποιο ωφέλη. Και εφόσον η δημοκρατία έχει πλεονεκτήματα, δεν είμαστε κατά. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το δημοκρατικό σύστημα για την αλλαγή της εξουσίας. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, οι μουσουλμάνοι εφάρμοσαν επανειλημμένα δημοκρατικές αρχές ή δημοκρατικά συστήματα. Και εγώ ως μουφτής και ως ύπατη θρησκευτική εξουσία στη χώρα μου θα ήθελα να επισημάνω ότι Ο Μουφτής ε, με βάση τα χαρακτηριστικά της θέσης του θα πρέπει πριν αναλάβει τα καθήκοντά του να έχει παρακολουθήσει σπουδές και να έχει ειδικευθεί σε θέμα ερμηνείας θρησκευτικών κειμένων με βάση θρησκευτικά κριτήρια. Αυτή είναι η μεθοδολογία της θεολογικής σχολής του Αλαζάρ και πρόκειται για μια μετριοπαθή ερμηνεία των θρησκευτικών κειμένων. Δεν ξέρω αν μας έχει μείνει χρόνος ακόμη. Όσον αφορά τους, ε, όσον τους ημάμιδες και ε, που λειτουργούν στα τζαμιά. Θέλουμε να διατηρήσουμε ένα διάλογο, γιατί κατά τη γνώμη μου ο διάλογος είναι απαραίτητος και αντιπροσωπεύει Μάλλον είναι αυτός που διευκολύνει τη συνεννόηση ανάμεσα στους λαούς. Πιστεύω να σας έδωσα απαντήσεις στις περισσότερες ερωτήσεις ε, που θέσατε. Σας ευχαριστώ που μου απευθύνατε τόσο κέρυες ε, ερωτήσεις που αντικατοπτρίζουν τη σοφία σας και την ε, τέλεια γνώση σας της κατάστασης στην Αίγυπτο και στον αραβικό κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. ich danke Ihnen sehr. Εξοχότατε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως και νομίζω ότι ήταν καλή αυτή η συνεδρίαση και αυτό θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά για την ε, διεξαγωγή καλού διαλόγου και πιστεύω ότι και ο ανοιχτός χαρακτήρας που επιδεικνύεται μας δείχνει ε, εδώ ότι αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η οδός για να συνεχίσουν οι συζητήσεις. Εξακολουθώ ωστόσο να πιστεύουν ότι οι τρεις μονοθεϊστικές ε, θρησκείες αν ε, ακολουθήσουν τα κοιτάπια τους θα έπρεπε και οι τρεις να είναι σε θέση να οργανωθούν με τρόπο λογικό η μία με τις άλλες. Γιατί καμία από τις τρεις αυτές τις θρησκείες δεν διακηρύσει το μίσος. Διακηρύσουν το Θεό της αγάπης και της συμφιλίωσης. Αυτή η ερμηνεία ή αν θέλετε το γεγονός, όπως είπατε, ότι η θρησκεία την χάνει εκμετάλλευση για άλλους σκοπούς είναι το πρόβλημα. Και αυτό ισχύει και για το Ισλάμ και για το χριστιανισμό και για τον Εβραϊσμό. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι μετριοπαθείς, οι οποίοι είναι άλλωστε και πλειονότητα και επιθυμούν την ειρηνική συνύπαρξη και είναι πραγματικά συντριπτική πλειονότητα και στις θρησκείες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά τη βία και για τη δική σας την περιοχή και για μας, ε, κοιτώντας ότι από τη χώρα μας έχουν φύγει 400 νεαροί άνδρες ε, και έχουν ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτος στη Συρία και στο Ιράκ και πολεμούν. Και απειλούν ότι θα έρθουν και σε εμά να κάνουν τα ίδια. Πάνω από 2.000 άτομα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και άτομα τα οποία δεν έχουν γυρίσει καν ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, σε ισλαμικές, ε, σε μουσουλμανικές οικογένειες, αλλά χριστιανοί που έχουν αλλαξοπιστήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και με τη δική σας προσπάθεια να προσπαθήσουμε κι εμείς να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση.